Meine Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρωινή μας συνεδρίαση. Πολύ καλημέρα σας. Και για την Λιθουανική Προεδρία που έπρεπε να πούμε ότι χαιρετούμε και υπό τη μορφή του Υπουργού Εξωτερικού, Εξωτερικών και εγώ ο ίδιος την προηγούμενη Παρασκευή κιόλας ήμουνα στο Βίλνιος όπου είχαμε την ευκαιρία να έχουμε συζητήσεις μαζί του με τον Υπουργό Εξωτερικών και με την Πρόεδρο. Πρέπει να πω ότι είχα συγκινητικές στιγμές που έζησα. Επισκέφθηκα τη Βουλή, το Κοινοβούλιο και ακόμα κάθισα στο έδρανο του κυρίου Λαντσμπέργης. Αυτό αποτόλμησα και έκανα. Κάθισα στο έδρανο του κυρίου Λαντσμπέργης. Και με μεγάλο θαυμασμό έζησα ξανά και βίωσα πόσο θάρρος χρειαζόταν και πόσο θάρρος είχε ο συνάδελφος Λαντσμπέργης και οι φίλοι του τότε. Τον Ιανουάριο νομίζω 91 δεν ήτανε που <clears throat> αντιστάθηκαν και με μεγάλο κίνδυνο προσωπικό υπερασπίστηκαν επιτυχώς την ελευθερία της χώρας τους. Γι' αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά αυτούς τους ανθρώπους. Χαίρομαι κύριε Υπουργέ για το ότι είσαστε εδώ ανάμεσά μας σήμερα και θα σας παρακαλούσα ιδιαίτερα να συζητήσετε μαζί μας ε, τα θέματα της πολιτικής διεύρυνσης και της πολιτικής γειτονίας ώστε να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα διότι έχουμε συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Και ακριβώς εμείς μαζί σας, για αυτούς τους λόγους, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ στενή συνεργασία, όπως επιθυμούμε. Χαιρόμαστε γιατί με αυτή την ευκαιρία έχουμε ανάμεσά μας και μια αντιπροσωπεία <clears throat> της κοινή Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση του Κοινοβουλίου της Βοσνίας Ερζεγοβίνης Καλώς ήρθατε θερμά υπό την ηγεσία του, Προέδρου. Καλώς ήρθατε. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα πολύ ευγενικά σας λόγια και για την εισαγωγή αυτή. Με μεγάλη ευχαριστήση βρίσκομαι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και όντας μέλος του Κοινοβουλίου γνωρίζω τι σημαίνει και πόσο μεγαλώνει η σπουδαιότητά του. Ελπίζουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά μαζί σας, να μένουμε σε επαφή, να διαβουλευόμαστε. Αυτή είναι η προθέση η δική μου και της ομάδας μου. Μετά από αυτή σας την εισαγωγή να σας πω δύο λόγια για τις προτεραιότητες της Λιθουανικής Προεδρίας. Εν συντομία φυσικά, διότι υπόθηκε ότι έχουμε να πούμε και περισσότερα για ζητήματα διεύρυνσης και εταιρικής σχέσης. Αλλά για να ξεκινήσω να σας πω ότι στη Λιθουανία πιστεύουμε στη συνέχεια των πραγμάτων και θέλω να ευχαριστήσω την Ιρλανδική Προεδρία για το έργο της. Εμείς αναλάβαμε από αυτούς και θα συνεχίσουμε, θα επεκτείνουμε όσα ξεκίνησαν αυτοί. Και ειλικρινά αυτό αντικατοπτρίστε στο πρόγραμμα τρίο προεδριών μαζί με την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η Λιθουανία θα εστιαστεί στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασία. Και αναγνωρίζουμε τρει πυλώνε. Ε, η αξιοπιστία τη Ευρώπη, η ανάπτυξη της Ευρώπη. Αξιοπιστία σημαίνει ένα αξιόπιστο δημοσιονομικό σύστημα, δημοσιονομική πειθαρχία, νομισματική ένωση και η αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική όσον αφορά και τους πολίτες, γιατί αυτοί την αισθάνονται. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι το έτος των πολιτών και δεν πρέπει να παραμείνει μόνο ένα σλόγγαν. Πρέπει να θεωρήσουν οι πολίτες ότι το περιβάλλον είναι πιο αξιόπιστο εδώ. Δεν είναι απλό το καθήκον αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση η αξιοπιστία θα αποτελέσει κομμάτι τη ατζέντα μα. Η ανάπτυξη τη Ευρώπη, η αναπτυσσόμενη Ευρώπη, σχετίζεται με την ενιαία αγορά και την υλοποίησή τη, με εστίαση στη ψηφιακό θεματολόγιο, την καινοτομία, την έρευνα και σίγουρα τη δημιουργία θέσεων εργασία. Η απασχόληση σήμερα ε, βρίσκεται σε θλιβερή κατάσταση. Η ανεργία ανέρχεται σχεδόν στο 25% στην Ευρώπη. Είναι συγκλονιστική αυτή η αριθμή πρέπει να κάνουμε κάτι. Γι' αυτό σε ορισμένε χώρε ξεπερνά και το 50%. Δεν μα εκπλήσει λοιπόν ο αριθμό των συναντήσεων όπου συζητούνται αυτά τα ζητήματα. Πρόσφατα συζητήθηκε να αφιερωθούν κάποια κονδύλια για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Τώρα θα έχουμε 8 δισεκατομμύρια για αυτά τα προγράμματα, αλλά οι κυβερνήσει επίση πρέπει να αναλάβουν ευθύνη, πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Οι Βρυξέλλε δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα, απλά διευκολύνουν, προσθέτουν κάποιου πόρου, αλλά στην πραγματικότητα οι εθνικέ κυβερνήσει είναι εκείνε που θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη. Και μια ανοιχτή Ευρώπη, ο τρίτο πυλώνα. Η ανοιχτή Ευρώπη αφορά τι σχέσει με τι τρίτε χώρε, τη διεύρυνση, τι ε, διαδικασίε προσχώρηση, τι ε, συμφωνίε σύνδεση και τι εταιρικέ σχέσει. Αλλά να σα αναφέρω εν συντομία ότι υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες στο κοινοβούλιο, τις οποίες πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε στο κοινοβούλιο αυτό και που ενσωματώνουμε σε αυτούς τους τρεις πυλώνες. Αυτέ οι προτεραιότητες είναι σίγουρα Αυτό σχετίζεται με τον πυλώνα ανάπτυξης, η εσωτερική αγορά ενέργειας που αποφασίστηκε από τους ε, επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων μέχρι το 2014 να δεξάλψει των νήσων, των ενεργειακών νήσων και εμείς είμαστε μια ενεργειακή νήσος και δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Μετά από 23 χρόνια ανεξαρτησίας παραμένει αυτή η κατάσταση αλλά αυτό δεν είναι πονοκέφαλο μόνο για εμά. Η ενέργεια είναι πονοκέφαλο και προτεραιότητα για πολλού από του συναδέλφου μα. Σίγουρα λοιπόν θα αποτελέσει κομμάτι του πυλώνα ανάπτυξη τη Ευρώπη και η μακροπεριφερειακή στρατηγική επίση για τις διαφορε χώρε και τη συνεργασία μαζί τους. Ε, έχουμε πολύ σημαντικούς οριζόντους δεσμούς με τις διάφορες χώρες, όχι μόνο συνεργασία, αλλά και πτυχές ε, ολοκλήρωσης με αυτές τις χώρες που θα λάβουμε υπόψη στις διάφορες αποφάσεις μας και δύο διεθνικού χαρακτήρα πυλώνες, εθνικές προτεραιότητες θα συμπεριληφθούν στον πυλώνα ανοιχτής Ευρώπης η ανατολική εταιρική σχέση σίγουρα αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις γι' αυτό αργότερα θα χαρώ να σας απαντήσω και να σας το περιγράψω περαιτέρω. Και η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης αποτελεί επίσης πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Έχουμε 650 χιλιόμετρα σύνορα με την Λευκορωσία και έχουμε κάποια εμπειρία από αυτό την οποία ευχαριστώ να μοιραστούμε μαζί σας. Τώρα όσον αφορά τη διεύρυνση, εμείς πιστεύουμε ότι ως Προεδρία θα πρέπει να είμαστε σίγουρα αμερόληπτοι ειλικρινείς διαμεσολάβητες και όχι να παίρνουμε ε, το μέρος του ενός ή του άλλου. Θα είμαστε προενεργοί, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους εταίρους να αναπτύξουν το θεματολόγιο με τον πιο θετικό δυνατό τρόπο χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της ουδετερότητας. Θα είμαστε θετικά επικοδομητικοί. Τρία μπλοκ θα ήθελα να αναφέρω σε αυτή τη διαδικασία διεύρυνση πρώτον η Ισλανδία. Συζητάμε τι αποφάσει εδώ και πολύ καιρό. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει. Γνωρίζουμε τώρα τη νέα απόφαση τη Ισλανδική κυβέρνηση. Πρέπει να τη σεβαστούμε. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί σα την εμπειρία μου. Πρόσφατα συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών ε, τη Ισλανδία, τον νέο Υπουργό, και είπε ότι αυτό πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το κλίμα διαλόγου. Πρέπει να διατηρήσουμε ό,τι κερδίσαμε κατά τη διάρκεια του διαλόγου τα τελευταία χρόνια με την Ισλανδία. Ακόμα και αν αυτή η κυβέρνηση δεν προωθήσει την ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρώπη, εμείς πρέπει να το σεβαστούμε και ας μείνουμε σε επαφή με την Ισλανδία, που είναι πολύ σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άλλο μπλοκ είναι η Τουρκία. Όλοι συζητούν για την Τουρκία και στις ειδήσει καθημερινά. Ήταν πολύ καλή απόφαση να ανοίξουμε το κεφάλαιο 22, πιστεύω, Ταυτόχρονα η επίβλεψη της κατάστασης, η παρακολούθηση της κατάστασης, μερικές φορές κάποιες ειδήσει μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας. Η διαδικασία η ίδια πιστεύω βοηθά να επηρεαστεί η κατάσταση επιτόπου. Εγγενώς πιστεύω δημιουργεί κάποια διαφορά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο, ο οποίος δεν είναι εύκολος, κρατάει πολύ, όπως όλοι γνωρίζουμε, παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό. και μετά τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια επίσης ε, είναι κομμάτι του παιχνιδιού τροποντινά την και εκεί θα πρέπει να είμαστε θετικά επικοδομητικοί για να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να προχωρήσουν, να προοδεύσουν και με μεγάλη μας ευχαρίστηση είδαμε την απόφαση έναρξης των συζητήσεων προσχώρησης με τη Σερβία. Ελπίζουμε ότι θα γίνει κατά την Προεδρία μας. Γνωρίζουμε τις συνθήκες, ξέρουμε πόσο δύσκολη ήταν η συμφωνία αυτή μεταξύ Κωσυφοπηδίου και Σερβίας Ξέρουμε πόσο δύσκολο ήταν για αυτούς, ε, ίσως και εις βάρος της ε, δημοτικότητας των κυβερνήσεων αυτών, αλλά ήταν μια στρατηγική απόφαση και πολύ σημαντικό τώρα είναι να υλοποιηθεί. Και θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να υλοποιήσουν αυτή την απόφαση, παρακολουθώντας στενά τη διαδικασία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με θετικό μάτι. Το ίδιο με το κοσυφοπαίδιο. Τις συζητήσεις ε, σύνδεσης θα τις ξεκινήσουμε σύντομα με θετικό πνεύμα. Εγώ πρόκειται να επισκεφθώ σε δύο εβδομάδε την περιοχή αυτή. Θα συναντηθώ με του ηγέτε, όπω και χθε με τον Πρωθυπουργό τη ΦΥΡΟΜ. Ε, συζητήσαμε λεπτομερώ τη δική του περίπτωση. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειε. Όλοι γνωρίζουμε την περίπτωση αυτή. Προβληματικέ σχέσει στην περιοχή, διμερεί σχέσει ε, προβληματικέ. Και όσον αφορά την υλοποίηση τη συμφωνία τη 1η Μαρτίου μετά από την κρίση πέρυσι. Αλλά έχουν τη δική του στρατηγική, μια θετική στάση Αναμφίβολα θα ήθελα να συνεχίσουν αυτή, σε αυτή την οδό ένταξης και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους βοηθήσουμε ως Προεδρία. Και διμερός, διότι έχουμε κάποια κοινά πράγματα, ιστορικές αποστολές για παράδειγμα, έχουμε πολύ καλή εμπειρία σε ορισμένες χώρες. Το είπα χθε στον Πρωθυπουργό, μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους και τη δική μας εμπειρία το Μαυροβούνιο. Επίσης ε, πρόσφατα πριν από μια εβδομάδα συναντήθηκα με τον Υπουργό Εξωτερικών όπου συζητήσαμε όλο αυτό το θεματολόγιο λεπτομέρως. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε τα πράγματα. Μια πιο δύσκολη κατάσταση είναι αυτή της Αλβανίας και της Βοσνίας Αρζεγοβίνης. Πριν από μια εβδομάδα η Αλβανία δοκιμάστηκε με τις εκλογές και τώρα τους ενθαρρύνουμε για μια ομαλή μετάβαση προς την κατάσταση, προς την ιδιότητα υποψήφιας χώρας. Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Αλλά ας διατηρήσουμε ανοιχτό αυτό το διάλογο. Το ίδιο και όσον αφορά τη Βοσνία. Δεν είναι εύκολη, περίπλοκη, μάλλον δύσκολη κατάσταση δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή, μια χώρα η οποία έχει μείνει πίσω στο ατζέντα ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι αποφάσει θα πρέπει να προέλθουν ε, από μέσα από τη χώρα βάσει της αρχής ε, ιδιοκτησίας ε, δεν μπορεί να είναι εντολές, να βασίζεται σε εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πολιτική ενότητα λοιπόν όλο αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να προωθήσουμε στους φίλους μας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Πολλά άλλα θέματα έχουν συμπεριληφθεί στην ατζέντα μου ζητήθηκε όμως να μην μιλήσω, να με ακρηγορήσω, οπότε μπορώ να δώσω απαντήσεις σε κάποιες ε, ερωτήσεις. Βλέπουμε τι συμβαίνει τώρα στην Αίγυπτο αυτές τις μέρες. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να παρακολουθούμε, να αναλύουμε την κατάσταση, να παρακολουθούμε τις ευθύνες μας γνωρίζοντας ότι η κοινωνία στην Αίγυπτο είναι διχασμένη και είναι βαθύ το χάσμα αυτό μεταξύ των δύο μέρων της κοινωνίας και είναι πολύ δύσκολο να αποφευθεί η διένεξη. Αλλά θα πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση αναλαμβάνοντας πλήρως τις ευθύνες. Και καλό θα είναι να παρουσιάσουμε σαφείς θέσεις και εμείς νομίζω στο Συμβουλίο προς τα τέλη του μήνα θα συζητηθεί η θέση μας όταν η κατάσταση θα έχει κάπως οριμάσει προτιμώ να δοθεί αυτό το μήνυμα νωρίτερα παρά αργότερα, για να το πω με ειλικρίνεια. Έχουμε και άλλα θέματα εντατικής συνεργασίας και Σήμερα αργότερα θα συζητήσουμε σε τριμερή διάλογο τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Πολύ δύσκολο θέμα, αλλά αρχίζει να υπάρχει σύγκληση απόψεων και ελπίζω ότι στην... η επόμενη φάση μπορεί να λάβει χώρα ακόμα και ενδεχομένω απόψε το βράδυ και ελπίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη σύγκληση. Δεν θα καλύψω όλα τα θέματα για να μην ε, σπαταλήσω και πολύ από το χρόνο σας και να μην γίνω βαρετός, αλλά με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος Σαλαφράνκα πρώτος που θα παρέμβει παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εξ ονόματος του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για την περίοδο της Προεδρίας σας για τους έξι αυτούς μήνες. Έχουμε πράγματι δυσκολίες σαν συνέπεια της κρίσης, αλλά βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή. Εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στα χρηματοοικονομικά μέσα και μας ανησυχεί ότι στον προϋπολογισμό για το 2014 για του χρόνου υπάρχει σημαντική περικοπή όσον αφορά την πρόταση, αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τα εξωτερικά θέματα και τη διεύρυνση, Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Τουρκία. Αληθεύει ότι είχαμε μια απόφαση αρχής ε, από το Συμβούλιο Υπουργών για το άνοιγμα του κεφαλαίου 22 υπό κάποιους όρους. Θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό το εγχείρημα να συμμετάσχει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτική γειτονία, για τις προσδοκίες που έχετε εσείς σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής του Βίνιους. Και πώς βλέπετε, πώς επικεντρώνεστε σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής. Με ενδιαφέρει πώς προσεγγίζει η Προεδρία σας κυρίως την Συμφωνία εταιρική σχέσης με την Ουκρανία λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η πρώην Πρωθυπουργό κυρία Τιμοσένκο και να μας πείτε πώς βλέπετε το θέμα της Συρίας και τις διαδικασίες διαβουλεύσεων Γενέβης 2 και πραγματικά με πολύ προσοχή παρακολουθούμε και την κατάσταση στην Αίγυπτο για την οποία κατάσταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια. Θα πρέπει επίσης να πούμε κύριε Υπουργέ και θα ήθελα κάτι να μας πείτε γι' αυτό για τις διαπραγματεύσεις ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και τι αναμένετε να πετύχετε εσείς κατά τη διάρκεια της δικής σας εξάμηνης προεδρίας. Και ολοκληρώνω με το τελευταίο να ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ για το ότι δεν ξεχνάτε και να μην ξεχνάτε και δεν ξεχνάτε τις σχέσεις με την Λατινική Αμερική και την επόμενη εβδομάδα στο Βίνιους ε, την την ε, κοινοβουλευτική συνέλευση ευρωλάτα ε, και όχι μόνο για την ε, φιλοξενία αλλά και για το ότι διάφοροι υπουργοί συμμετέχουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούστηκε η παρέμβαση. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που είσαστε εδώ. Τις καλύτερες επιτυχίες, ευχές μας για την επιτυχία της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για την δική σας προσέγγιση προς την Λευκορωσία, Μπέλαρους. Σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική έκθεση για την ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Μπέλαρους ε, που τίθεται υπό έγκριση, υποψήφιση και έγκριση. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις επ' αυτού. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μια ερώτηση που κάποιοι και τουλάχιστον από τη χώρα μου μου έθεσαν ως ερώτημα. Είναι νομίζω σημαντικό το ερώτημα αυτό. Έχω μια απάντηση εγώ, αλλά θέλω τη δική σας απάντηση ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση το πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Το ενέκρινε αυτό το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Αίγυπτο. Και η άλλη μου ερώτηση είναι πώς εσείς αντιμετωπίζετε εξ ονόματος της Προεδρίας, πώς βλέπετε την οδό. Κάποια από τα κράτη-μέλη έδρασαν με αυτό το συμβάν που σημειώθηκε με το αεροπλάνο του Προέδρου της Βολιβίας Εύω Μοράλες παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο αναγκάζοντάς το να προσγειωθεί. Δεν νομίζετε ότι το να μην υπάρχει προστασία για κάποιον ο οποίος κατήγγειλε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου ε, όσον αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών, ότι και αυτό είναι μια παραβίαση δικαίου. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, έκλεισε ο κατάλογος των αγορητών. Και δεν θα μπορέσουν και όλοι νομίζω φοβάμαι να παρέμβουν, διότι πιέζει πολύ ο χρόνος και είναι πολύ, μεγάλη, ε, πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Αν το δυνατόν περισσότεροι θέλουν να ενταχθούν σε αυτόν τον κατάλογο, τότε το πολύ 1,5 λεπτό θα παρεμβαίνετε. Συμφωνείτε λοιπόν, παρακαλώ να τηρείτε το όριο του 1,5 λεπτού, γιατί πιέζει ο χρόνος. Ο κύριος Σακασί, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την Προεδρία σας. Ελπίζουμε ότι θα είσαστε ε, ιδιαίτερα φιλόδοξοι στις προσπάθειές σας ε, να κάνετε τόσες αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την διεύρυνση και να ξεκινήσω με την Τουρκία πιστεύω, αλλά και άλλοι στην Άλντε πιστεύουμε, ότι το κεφάλαιο 23 είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ζητήσω, να, όχι να είστε θαραλέος, γενναίος, αλλά φιλόδοξος όσον αφορά το άνοιγμα και άλλων κεφαλαίων, διότι αυτό θα είναι προς όφελος και των κατοίκων της Τουρκίας, αλλά της περιοχής γενικότερα και της Ευρώπης, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά κάποιες ιδιαίτερες χώρες, αναφερθήκατε στην Βοσνία. Ευτυχώς η αντιπροσωπεία της Βοσνίας από το Κοινοβούλιο είναι εδώ σήμερα και θα συζητήσουμε αργότερα τι θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε. Η, ε, η προσχώρηση της Κροατίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Από την 1η Ιουλίου θα υπάρχει αλλαγή στις εξαγωγές από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Επομένως πρέπει να γίνει κάτι έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές αλλά και να ξεπεράσουμε κάποιες ε, συνέπειες. Ε, θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να τις βοηθήσει, να βοηθήσει για να ξεπεραστούν ε, τα προβλήματα. Ευχαριστώ τον Υπουργό, ευχαριστώ τον Πρόεδρο καταρχά και τον Υπουργό που ήρθε. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για το Σύνοδο Κορυφής στο Βίλνιους. Στην προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής θεωρείτε ότι πρέπει να ε, προετοιμαστείτε ε, έτσι ώστε να συζητήσετε καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θα γίνει μετά την σύνοδο του Βίλνιους, ποιες είναι οι εξελίξεις που προβλέπετε ή τέλο πάντων ε, θεωρείτε ότι μετά την σύνοδο θα υπάρχουν εξελίξεις με τις χώρες τις ανατολικές Ανατολικής Γειτνίας. Σας ευχαριστώ και Πρόεδρε και ευχαριστώ τον Υπουργό ε, για το Σύνοδο, ε, για το Βίλνιους, ε, Γεωργία, Αρμενία και Μολδαβία. Έχετε να μας πείτε κάτι, υπάρχουν και σε κάποιες χώρες προεδρικές εκλογές που θα γίνουν. Υπάρχουν και συμφωνίες συνεργασίας τι θα γίνει αν κάποιες χώρες γίνουν δεκτές και η Ουκρανία απορριφθεί. Αυτό πώς θα δικαιολογηθεί εάν απορρίψουμε την Ουκρανία, πώς θα βοηθήσουμε την κυρία Τιμοσέγκο που βρίσκεται στη φυλακή για την ε, Λευκορωσία και άλλοι συνάδελφοι το ανέφερα και το έχουμε εδώ. Αλλά αυτή η πολιτική του καρότου και του ραβδιού λειτουργεί με το καθεστώς του Λουκασέγκο και για τα Δυτικά Βαλκάνια, επειδή είμαι και εισηγητής για το Μαυροβούνιο, δεν χρειάζεται να σχολιάσετε για το Μαυροβούνιο, αλλά για τις συζητήσεις Σερβίας Κωσυφοπεδίου και πώς διαμορφώνεται το μέλλον του Κωσυφοπεδίου. Επίσης το όνομα του ονόματος της Μακεδονίας, πώς ε, θα μπορέσουμε να επιτρέψουμε στην Μακεδονία να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρησή της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Ήθελα να αναφέρω μόνο ένα πράγμα, η διαδικασία διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάδια, η χώρα σας ανέλαβε την Προεδρία σε καλή στιγμή για να συμβάλλει στη διαδικασία. Διότι κοιτώντας την κατάσταση εκεί αυτή τη στιγμή είναι πολύ θετικό σήμα αυτός ο αρελισμός, αυτή η ρεαλιστική προσέγγιση που μας ε, δείξατε στην εισαγωγή σας. Εγώ συμφωνώ. Η ιστορική συμφωνία Σερβίας και Κωσυφοπεδίου οθεί τα πράγματα προς τα εμπρός και μετά τις εκλογές ε, στην Αλβανία η μετάβαση της εξουσίας προς το παρόν φαίνεται να πηγαίνει καλά. Όλοι οι πολιτικοί ηγέτες τα λένε όλα σωστά. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή ρεαλιστική προσδοκία σύντομα για τη χώρα αυτή. Το μόνο σχόλιο που έχω να πω, έχουμε του συναδέλφου εδώ από τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, ξεκινήσαμε χθε τι συζητήσει και του προσθέσουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση και ξέρουν τα προβλήματα, ξέρουμε και εμεί ποια είναι τα προβλήματα, αλλά χρειαζόμαστε αποτελέσματα και όλοι γνωρίζουμε πώ μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτό. Εσείς αναφέρατε και αυτό ότι πρέπει να είστε προενεργοί και φιλόδοξοι σε αυτή τη διαδικασία. Και συμφωνώ με αυτό διότι η Σερβία θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο μόλις, αλλά μην περιμένουμε μέχρι τότε. Έχουμε πολλά να κάνουμε στο μεταξύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε και καλή τύχη. Ό,τι καλύτερο για την Προεδρία σας. Αναφέρατε τη διαδικασία διεύρυνσης. Θα ήθελα να τονίσω όταν μιλάμε για την Τουρκία ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους μου Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στο κεφάλαιο 23. Αυτό που είναι κρίσιμο στην Τουρκία είναι ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μια φάση εκπόνησης ενός νέου συντάγματος και αυτό είναι κρίσιμη σημασία. Εάν καταφέρουν οι Τούρκοι να αποκτήσουν ένα φιλελεύθερο, δημοκρατικό, δυτικού τύπου σύνταγμα με ε, σωστή, ε, ε, σωστό καταμερισμό των εξουσιών. Αυτό θα είναι πολύ καλό σήμα και θα βοηθήσει την όλη διαδικασία. Όσον αφορά τη διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια, δεν έχω ιδιαίτερε αμφιβολίε για την Αλβανία. Παρατηρήσαμε τις εκλογές, έκαναν τεράστια πρόοδο, ήταν οι καλύτερες εκλογές ποτέ όσον αφορά τι συμπεριφορέ των κομμάτων, τα οποία συνεργάζονται μεταξύ του. Α δούμε λοιπόν πώ θα που θα καταλήξει μεταβατική αυτή περίοδος και πιστεύω ότι μετά μπορούμε να πιέσουμε για το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Εμείς δεν κάνουμε διαφορά μεταξύ Σλάβων και μη Σλάβων στα Δυτικά Βαλκάνια. Να κάνω μια ερώτηση για τη Λευκορωσία. Αναφέρατε την ενέργεια. Πώς βλέπετε την ε, εταιρική σχέση σε θέματα ενέργειας με τους γειτονές σας στη Λευκορωσία και μετά τίθεται και το ερώτημα της ασφάλειας της πυρηνικής ενώ ασφάλειας των πυρηνικών ε, εργοστασίων που χτίζονται στη Λευκορωσία. Τι θα κάνουμε γι' αυτό ώστε να μπορούμε να έχουμε και κάποια αποτελέσματα για να επιληθεί το ζήτημα της ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λιθουανία έχουν κοινέ πολιτικές προτεραιότητες. Μεταξύ αυτών η ανατολική γειτονία, αυτή η σχέση από την οποία έχουμε προσδοκίες μέσα από τις πρόοδους που επιθυμούμε να σημειωθούν. Πρώτο ερώτημα. Αυτό το επίπεδο των κοινών προτεραιοτήτων από κοινού μετράται και αξιολογείται από την Λιθουανία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμιά φορά στο λιθουανικό τύπο ασκούνται επικρίσεις σαν μόνο η Λιθουανία λέει να θέλει να εμφανιστεί πολύ καλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αν δεν συμβαίνει αυτό τότε δεν συμβαίνει και τίποτα τρομερό. Πρόοδος λοιπόν και προαγωγή αυτού του θέματος που είναι σημαντική υπόθεση για τους συνδεδεμένους εταιρούς υποσχέσεις σύνδεσης αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λιθουανία θα μπορούσε ως διαμεσολαβητής να δράσει μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα, η προσέγγιση αυτή στην Λιθουανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποια είναι. Με τον ίδιο τρόπο μετράτε και αξιολογείτε ή είναι διαφορετικές οι διαδικασίες. Αν εμείς τη δική μας πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αν θυμηθούμε ποια ήταν η πορεία μας μέχρι να ενταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια τεχνητά προβλήματα δημιουργήθηκαν και υπήρξαν ως προς τότε δηλαδή η βαλτική προσέγγιση, η προσέγγιση των βαλτικών χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρισκόταν λέει ε, ενάντια στα συμφέροντα της Ρωσίας. Τότε οι ευρωπαϊκές δομές και οι δομές του ΝΑΤΟ δεν απέκρυψαν τα πράγματα και είπαν πως είχαν. Τώρα τι συμβαίνει σήμερα ακριβώς μπορεί μια ελεύθερη απόφαση να απορρέψει για τέτοια θέματα σαν απόφαση εναντίον κάποιου. Μπορεί να ερμηνευτεί έτσι ενδεχόμενα. Θα ήθελα να αναφέρω ότι στη γενεοδορία μας δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιθώρια. Σε ευχαριστούμε πολλά πολύ. Ο κύριος Υπουργός έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά. Όπως αναμένεται, το θέμα της εταιρικής σχέσης είναι εκείνο το οποίο συχνότερα αναφέρθηκε στις περισσότερες πτυχές και θα παραμείνω περισσότερο στις εξηγήσεις μου γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα για το ίδιο το γεγονός. Όταν με ρωτούν και συχνά με ρωτούν ποια θα μπορούσε να είναι η επιτυχία της εταιρικής σχέσης και σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφής, ενδιαφέρον το ερώτημα και σε σχέση με το ίδιο το ε, πρόγραμμα πρόγραμμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι ε, φιλοδοξίε μα και τι προσδοκίε μα που πολλέ φορέ μπορεί να βρίσκονται σε πολύ ψηλό επίπεδο και μετά να υπάρξουν απογοητεύσει. Αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι σωστό ούτε για του εταίρου αλλά ούτε και για μας. Διότι το ίδιο το γεγονό ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέταξαν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη τη Συνόδου κορυφή είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Λοιπόν, για αυτό το θέμα ε, σε σχέση με τη Σύνοδο Κορυφή, ε, θα είναι ο σεβασμό ακριβώ για αυτό το θέμα θέμα και αυτό αποτελεί μέρος της επιτυχίας και το να μπορέσουμε μετά τη Σύνοδο Κορυφής να πούμε ότι έχουμε μια στρατηγική για την ε, ε, πολιτική γειτονία έναντι των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης να υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα more for more να ωφεληθούν περισσότερο αμφότερες οι πλευρές καμιά φορά ακούγονται ωραία αυτά αλλά πρέπει να υλοποιούνται αυτά more for more σημαίνει και πρέπει να σημαίνει κάτι χειροπιαστό να υπάρχουν αυτά αποτελέσματα και να υπάρχουν μηχανισμοί για να επιτευχθούν αυτά και ουσιαστικά αναφερθήκατε και για την προοπτική και μετά το 2013. Πρέπει να υπάρχει ένα όραμα μέσα σε αυτή την προοπτική. Δεν τερματίζεται η ζωή με αυτή τη σύνοδο ξεκινά μόνο και μετά το 2013 είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει. Τούτων λεχθέντων και πάλι πρέπει να πω ότι μια και αναλώνουμε μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό είναι νόμιμο και θεμητό συζητώντα θέματα τα οποία είναι φλέγοντα θέματα, Συρία, Μάλι και πολλέ φορέ και μέχρι τα μεσάνυχτα και πρωινέ ώρε. Και αυτό είναι νομιμο νομιμοποιημένο και θεμητό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας παγκόσμιος παίκτη σε αυτή τη σκηνή, στην παγκόσμια κονίστρα. Σίγουρα έχουν αυτά τα πράγματα τη σημασία τους, αλλά μην ξεχνάμε το όραμα για την Ευρώπη ελεύθερη και μεγάλη που δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Να μην νομίζουμε ότι επειδή δεν υπάρχουν ε, σειράξεις και συγκρούσεις ε, όλα πάνε καλά. Πολλά θα πρέπει να γίνονται αναθεωρήσεις, αξιολογήσεις σε τακτά διαστήματα για να μπορούμε να ε, σημειώσουμε επιτυχίε. Μια πρόσθετη θα μπορούσε να είναι και κάποιοι ρώτησαν κιόλα ε, σε σχέση με την εξοικείωσή τους και γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες αυτών των κατοφυλακίων την ε, υπογραφή συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ουκρανία σε αυτή τη σύνοδο κορυφής. Είναι δυνατόν, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αποστέλουμε μηνύματα ότι ε, διαδραματίζονται όλα αυτά στο ίδιο πεδίο δράσης. Είναι επικοδομητική και η αποστολή του Κοινοβουλίου που απεστάλλει από τον πρόεδρο από, από πλευράς Προεδρίας ήταν πολύ επικοδομητικό να υπάρχει αυτό το θετικό κλίμα. Και όταν έχουμε και διμερείς επαφές, όταν πηγαίνουμε με ομάδες ε, και είναι χρήσιμο και αυτό και μπορώ να αναφέρω και το παράδειγμα, όταν πήγα ο ίδιος ε, και με τον κύριο Σικόσκι, Υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας και με τον κύριο Τίμερμανς, Υπουργό από την Ολλανδία και από πλευράς ε, της Δανίας με Υπουργό. Πήγαμε στο Κίεβο, συναντήσαμε τον Γιαννουκόβιτ, συζητήσαμε αυτά τα θέματα. Είναι ένα υπόδειγμα πώς θα πρέπει να γίνονται από όλους μας αυτά. Επιλέξαμε τρεις τομείς. Φυσικά πολλά περισσότερα περισσότερα μπορούν να γίνουν. Είπαμε στους Ουκρανούς, σε τρεις άξονες πρέπει να δώσετε χειροπιαστά αποτελέσματα. Ένα σύστημα για τις εκλογές, για να επιτευχθούν ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές, εποπτεία. Υπάρχουν μηνύματα ότι έχει σημειωθεί πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, παρόλες ελλείψεις, πράγμα το οποίο δεν μας εκλείσει. αλλά χρειαζόμαστε τέτοιου είδους θετικές ειδήσει από την Ουκρανία. Και εκεί είναι ένας τομέας όπου μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες προόδου επ' αυτού. Δεύτερον, δικαστική ουσιαστική μεταρρύθμιση εν τέλει. Δεν πάει όσο γρήγορα όσο θα θέλαμε. Είναι πολύ ευαίσθητο, υπερβολικά ευαίσθητο αυτό το θέμα για αυτούς. Αλλά είναι καλά τα μαντάτα, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν χειροπιαστά. Δεν λέμε απλά και μόνο να υπάρξουν βελτιώσει. ξέρουν ακριβώ τι πρέπει να βελτιωθεί, με ποια νομοθετήματα, ποιου νόμου που πρέπει να εγκριθούν. Είναι μια σφαιρική ε, διαδικασία ολοκληρωμένη. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ε, και η δράση του ε, δημόσιου εισαγγελέα, του κρατικού εισαγγελέα, εκτό πολιτικού ελέγχου, ε, πολιτιακού ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχουν τα ειχέγγυα για την ανεξαρτησία λοιπόν της δικαιοσύνης και της μεταρρύθμισης στον δικαστικό τομέα. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς αυτός των δικαστικών ε, θεμάτων και των μεταρρυθμίσεων. Και το θέμα λοιπόν ε, το της επιλεκτικής δικαιοσύνης. Όσοι παρακολουθούν τα πράγματα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται με την Γιούλια Τιμοσέγκο. Και όλοι αυτοί γνωρίζετε συνάδελφοι τι γίνεται. Μπορεί να μην αρέσει ή να το βρίσκεται περίεργο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η, δοκιμασία, η λιδία λίθος, λίθος για το κράτος δικαίου και την ένωμη τάξη. Αν δεν γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές υπάρχουν προβλήματα, πρέπει να επιληθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα προσκόμματα και εμπόδια. Όλα αυτά τα οποία παρακολύουν ε, την ελεύθερη δικαιοσύνη και λειτουργεί μια επιλεκτική δικαιοσύνη. Το βλέπουμε αυτό το τι έγινε με την Τιμοσέγκο. Χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Και θα ήταν μια ανθρωπιστική, α το πούμε έτσι, ε, παρέμβαση. Δεν θα ήταν κάτι το οποίο θα έβλαπτε το πολιτικό σύστημα. Θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται αυτό, να τη παρασχεθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε αυτά και να ολοκληρωθεί η πορεία των Ουκρανών προ αυτού του στόχου. Καθότι γνωρίζουμε λοιπόν, είναι πολύ επικοδομητική η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, διότι τρέχει ο χρόνο και δεν μα παρέχει ευκαιρίε, ε, δεν μα δίνει διάλειμμα προς ε, δική μας, ε, ε, δικό μας προβληματισμό και δράση. Να περιμένουμε μέχρι ότου καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Όχι, δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να δράσουμε ταχύτατα. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι και, πρέπει, και το γνωρίζουν κιόλα αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει περίοδος αναμονής και διαλύματος. Αν συμφωνείτε μαζί μου, η περίπτωση της Ουκρανίας δεν είναι μια άλλη περαιτέρω τεχνική συζήτηση με άλλη μια χώρα για οικονομική ολοκλήρωση, εταιρική σχέση. Όχι, είναι μια γεωπολιτική σημασία και σπουδαιότητα Στη διαδικασία. Δηλαδή δείχνει και κατά πόσο θα μπορέσουμε να, είμαι, να είμαστε επιτυχείς με το πρόγραμμά μας ε, για την Ευρώπη. Λιγότερο επιτυχής για παράδειγμα ή περισσότερο επιτυχής. Να τα σκεφτούμε αυτά. Αυτές είναι οι ευθύνες μας. Δεν λέω να τα κάνουμε εις βάρος των απαιτήσεών μας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω πρέπει ως γεωπολιτική σπουδαιότητας διαδικασία να το αντιμετωπίσουμε, να μην βρεθούμε και βρεθούν στην πλευρά των χαμένων ε, εκείνων που έχασαν το παιχνίδι. Αυτό το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη. Για τις υπόλοιπες χώρες. Να πω, για αυτές τις έξι χώρες που είναι χώρες μέλη της ανατολικής ε, γειτονικής σχέσης ε, είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν μπορούν ε, να, υπα... ακολουθήσουν ένα κοινό πρότυπο ισοπεδωτικά σε σχέση με άλλες χώρες. Κάνουμε λόγο για την Ουκρανία, δυνατότητα να υπογραφεί η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης για παράδειγμα με αυτήν. Άλλες χώρες έχουν διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα για να μπορέσει να προαχθεί και για τη Μολδοβία, για παράδειγμα, Μολδόβα που εξήλθε από την και που αντιμετώπισαν την κρίση και επέλυσαν το θέμα με την κυβέρνηση δεν έχασαν χρόνο. Ο, προχώρησαν στις διαπραγματεύσεις προς την ολοκλήρωσή τους και αυτό ήταν ένα και εκτιμένο. Τώρα που μιλάμε και καθώς μιλάμε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και με τη Γεωργία. Κάνω λόγο για το τεχνικό σκέλος αυτού του θέματος. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν και προηγούμενα για τη διαδικασία συμβίωσης, συνύπαρξης μεταξύ Προέδρου και κυβέρνησης, ε, μεταξύ του διαλόγου δηλαδή ε, κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Το ίδιο μήνυμα είναι εκείνο το οποίο αποστέλουμε προς τους Γεωργιανούς. Να τους πούμε πρέπει να συμμορφωθούν και να ε, μπορέσουν να φερθούν σωστά. Δεν μπορούν να φυλακίζονται οι πρόσωποι της αντιπολίτευσης. Και φυσικά εδώ πρέπει να σεβαστούν και να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη όλα αυτά. Αυτά είναι τα μηνύματα που αποστέλουμε προς την Γεωργία. Δεν είναι πάντα πολύ επικοδομητικά για την ε, κατάσταση, δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται όταν γίνονται τέτοιες επιπλήξεις, αλλά σίγουρα μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσουμε να προγάγουμε τα θέματα. Και με την Αρμενία το ίδιο. Μπορούμε να το, κάνουμε, να μπορούμε να το προχωρήσουν αυτό και αυτό το μήνα. Όσοι υλοποιήσουν αυτές τις προϋποθέσεις θα μπορέσουν να προχωρήσουν παραπέρα. Το θέμα λοιπόν ε, για τη Σύνοδο Κορυφή ε, και το χρονικό διάστημα που απομένει είναι κάτι το εφικτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι περνάει από το χέρι δείκτης για να ανταποκριθούμε στι προσδοκίε και πρέπει να υπάρξουν και περαιτέρω επιτυχίε πέρα από τι επιτυχίε που ανέφερα πιο πριν στην έναρξη του λόγου που, με τον οποίο σα προσφώνησα και τον διάλογο για τι θεωρήσει διαβατηρίων. Ε, δεν θέλω τώρα να το συζητήσω αυτό μαζί σα, αλλά ε, ε, ε εκ περιτροπή πρέπει να συζητείτε. Δεν είναι μόνο το όλο θέμα ε, και το μόνο όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και το ευρασιατικό όραμα, η τελωνιακή ένωση. Υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα από διάφορες πλευρές. Δεν θέλω να ε, οδηγηθούμε σε μια συγκρουσιακή λογική ότι αυτά όλα αντιμετωπίζουν με τοπικά το ένα ε, με το άλλο όσον αφορά αυτές τις προοπτικές για το μέλλον. Αλλά και πάλι με το θέμα παρατηρητών χωρίς παραβίαση κανόνων του υπενθυμίζουμε δεν μπορείτε να υπογράψετε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ευρώπη και μετά να έχετε μια ίδια συμφωνία όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση από πλευρά σας. Δεν μπορείτε να ε, κόψετε τις γέφυρες. Πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες του παιχνιδιού. Πρέπει να επιλέξετε με υπεύθυνο τρόπο, όχι εις βάρος σας το πω έτσι, της μακροπρόθεσμης στρατηγικής σας, θα μπορούσε να, είναι και μια πιο, να υπάρχουν και πιο βραχυπρόθεσμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πρέπει να επιλύσουν, αλλά μέσα στην τεράστια αγορά των 500 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανοίγει τεράστιες προοπτικές για αυτούς και μακροπρόθεσμα θα έχουν και κέρδη, θετικά κέρδη. Το να, ε, ατέρμο, με ατέρμονα τρόπο να συζητούν αυτά τα θέματα και να φτάνουν ε, στον τύπο. Δεν θα πάρουμε εμεί τι αποφάσει για, αυτά, για εσά. Εμεί ε, θα σεβαστούμε τι δικέ σα αποφάσει. Αλλά θα προτιμούσαμε παρόλα αυτά την ευρωπαϊκή πορεία. Μια κοινή σύγκληση στην πορεία ε, ε ημών και ημών, με ύψιλον και με ήττα ώστε να υπάρξει μια α το πω έτσι ομαλή πορεία. Τώρα, για την γεωργία όπω αναφέρθηκε πιο πριν, είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι ένα μαθηματικό υπολογισμό, α το πω έτσι, ω ένα άθροισμα και βασιζόμαστε σε αρχές, σε αξίες, ε, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην ένωμη τάξη, στο κράτος δικαίου. Οποιοδήποτε πράγμα παραβιάζεται πρέπει με σαφές μήνυμα που αποστέλουμε να ε, το καταγγέλουμε και να πούμε στους Γεωργιανούς ότι πρέπει να φτάσουν σε ένα σημείο όπου θα είναι ε, χωρίς επιστροφή, αμετάκλητη πλέον η πορεία τους υπέρ μιας τέτοιας ευρωπαϊκής προοπτικής και επιλογής. Για τον Κάφκασο και το Αζερμπαϊτζάν, πάλι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Το Αζερμπαϊτζάν δεν θα να είναι κράτος μέλος Ευρωπαϊκή Ένωση, Θα προσαρμόσουν οι Αζερμπαϊτζανοί το νομικό του σύστημα ε, προ αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν συνειδητοποιήσει και γνωρίζουμε ότι είναι ε, μεγάλο παίκτη για τα ενεργειακά θέματα. Μπορεί να είναι αδιάφοροι, μπορεί να είναι ουδέτεροι, μπορεί να είναι και επικοδομητικοί. Θετικά διακείμενοι υπέρ ημών στα ενεργειακά θέματα. Α συζητήσουμε λοιπόν, α διαβουλευτούμε, α έχουμε ένα διάλογο μαζί του. Είναι πολύ σημαντικό. Ρεαλιστικά πάλι και πραγματιστικά, χωρί ε, να αποβεί αυτό ει βάρο των δικών μα αρχών και αξιών διότι γνωρίζουμε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Ο πύχη όμω δεν θα τεθεί τόσο υψηλά ώστε να υπάρξουν προσκόμματα και δυσκολίε. Α σεβαστούμε λοιπόν αυτέ τι επιλογέ και α κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να διευκολύνουμε και να βελτιστοποιήσουμε τι δικέ μα ε, επιδόσει. Τώρα για τι άλλε χώρε. Μολδόβα, Μολδαβία ήδη την προανέφερα. Κατά τα άλλα γιατί η Μολδαβία είναι πολύ, ένα πολύ καλό παράδειγμα όταν έχουμε την εφαρμογή τη αρχή more for more. Περισσότερα για περισσότερα. Κάνουν πολλά όσον αφορά τι θεωρήσει διαβατηρία διαπραγματεύονται επιτυχώ και μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, να στεφθεί με επιτυχία μέχρι τα τέλη του έτου. Ε, τότε πρέπει λοιπόν να εξαιρεθούν από τι θεωρήσει διαβατηρίων, αν τα καταφέρουν. Αυτή είναι η εφαρμογή τη αρχή περισσότερα για περισσότερα. Αν κάνουν αυτά τα οποία εμεί προσδοκούμε και αναμένουμε, τότε πρέπει να ανταμυφθούν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερα προσκόμματα και δυσκολίε. Δεν είναι αυτή η αρχή περισσότερα για περισσότερα, more for more. Βλέποντα τι κάνει λοιπόν η Μολδόβα. Και τώρα για την Μπελαρού στη Λευκορωσία. Όταν κάθε κανεί εδώ και είναι άνετα, βρίσκεται άνετα ή και οι αποστάσει είναι μεγάλε. Για την Βίλνιου όμω έχουμε διαφορετική κατάσταση. 30 χιλιόμετρα είναι όλα και όλα η απόσταση μέχρι τα σύνορα και 40 χιλιόμετρα από εκεί που θα οικοδομήσουν, θα εγείρουν το νέο του πυρηνικό σταθμό με του πυρηνικού αντιδραστήρε. Υπάρχουν πολλέ ευαισθησίε λοιπόν και πάντα δίνουμε αυτό το παράδειγμα. Ζητώ συγγνώμη για την επανάληψη αυτών των παραδειγμάτων όταν το αναφέρω επανειλημμένα, τα αναφέρω αυτά επανειλημμένα. Η θέση μα είναι η ίδια όμω. Δεν έχει αλλάξει την τελευταία φορά από την οποία, σε κάτι την συναντηθήκαμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ δαπανηρό. Ε, μπορεί να γίνει αυτό και φθηνότερα, με, το ίμιση και όλα φθηνότερα. Και θα το κάνουν αυτό. Τι σημαίνει αυτό, να ε, ε, εγερθεί με φθηνότερο τρόπο σε σχέση με τον προϋπολογισμό που αρχικά είχε προϋπολογιστεί. Τα γνωρίζετε τι σημαίνουν αυτά και επανέρχομαι στι προτεραιότητε που ανέφερα στην αρχή. Δεν τα ανέφερα όλα αυτά λόγω του ότι πίεζε ο χρόνος. Και έχουμε εδώ και τα ενεργειακά θέματα και την ενεργειακή πολιτική. Είναι ένα από τα θέματα που στην Προεδρία μας θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Έκθεση ενεργειακής πρόοδου για την αγορά ενέργειας υποβολή έκθεσης πρόοδου σε ε, σχέδια και εγχειρήματα κοινού συμφέροντος που συνδέονται με την ενέργεια και εξωτερική ενεργειακή πολιτική και τα συμπεράσματα θα συζητηθούν επ' αυτού κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρία Τι σημαίνει εξωτερική πολιτική. Πρέπει να μιλάμε μια ενιαία φωνή η Ευρώπη για αυτά τα θέματα και αυτό είναι πολύ σοβαρό για όλους. Πιστεύω ότι ε, ο πυρηνικός αντιδραστήρας 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα αυτής της χώρας ε, με αμφισβητήσιμη ποιότητα αυτού του αντιδραστήρα δεν πρέπει να είναι μόνο δικό μα πονοκέφαλος και δική μα ανησυχία τώρα εδώ σε σχέση με διμερεί προβλήματα που μπορεί να έχουμε εμείς δεν θέλω εγώ να, τα, να προβληματίσω άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με τέτοιο εθνικό πονοκέφαλο. Όχι, πρέπει όμως με ευθύνη, με μία φωνή να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Για την οδηγία για παράδειγμα ασφάλειας πυρηνικών αντιδραστήρων, Nuclear Safety Directive και είναι κοινό αυτό το εγχείρημα και αυτή η πολιτική. Θα πρέπει να συνεργαστούμε. Έχουμε ήδη συλλέξει ε, πείρα και εμπειρία σε, αυτό, σε αυτά τα πεδία Επ' αυτού του θέματος θα ήθελα όλους σας να σας καλέσω να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε για να υπάρξει αυτή η επιτυχία αυτή της ενιαίας ενωμένης φωνής από την Ευρώπη και για την ανατολική ευρωπαϊκή γειτονική σχέση. Ας μην μακρηγορήσω τώρα. Είναι τόσο σημαντικά αυτά τα θέματα και τόσο ενδιαφέροντα που μπορεί κανείς να μακρηγορήσει. Υπάρχουν δύο θέματα λοιπόν. Το να περιμένει κανείς να δει το τι θα γίνει κατά το δοκούν ή η ενεργός ε, ε, ε θέση και δραστηριοποίηση. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναμείνουμε να δούμε το τι θα γίνει. Φυσικά είναι νόμιμα πολλά πράγματα και ε, φυσικά κάνουν λάθη κάποιοι και έχουν ε, ελλείψεις. Αλλά ας είμαστε θετικοί, ας δούμε το τι θα γίνει. Λακωνικότατα και τηλεγραφικά για την Τουρκία. Ναι, να, αν μπορούμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Αυτή η ε, διαδικασία προσχώρησης, ένταξης είναι θετικό να μπορέσει να συνεχιστεί. Και για το 22-23 κεφάλαια, το 19, το 17 κοινωνική πολιτική, μακάρι να μπορούσε να ανοίξει ε, τώρα για, τη, για την Αλβανία δεν έχω ε, επιφυλάξεις να προχωρήσει να αποκτήσει το καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας εντάξει να μπορέσουμε να το κάνουμε να υπάρξει μια ήπια χωρίς προβλήματα μετάβαση και ελπίζω ότι τα πολιτικά κόμματα θα είναι έτοιμα να υπομισθούν τις ευθύνε τους από τα κόμματα της Αλβανίας δεν έχω επιφυλάξεις έχω ε, μάλιστα μπορώ να πω ότι έχω θετικά διά, ε, έχω θετικές διαθέσεις έναντι της ε, ε, Αλβανίας. Τώρα, ένα λεπτό. Τι είπατε εσείς? Βοσνία, μάλιστα. Βοσνία. Σωστό. Όπως προανέφερα, αν θεωρήθηκε ότι είμαι επιφυλακτικός, ε, ε, όχι, είμαι ρεαλιστής. Θυμάμαι για τη Βοσνία. Είχα και κιόλα περάσει και ένα διάστημα στο ΝΑΤΟ και έχουμε συζητήσει εκτενώς αυτά τα θέματα και λεπτομερώς. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε σχέση με την χώρα αυτή να μπορέσει να είναι πιστική προσέγγιση αυτή ότι μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες της στο κρατικό επίπεδο αποτελεσματικά διότι διαφορετικά θα επανέρχονται τα ερωτήματα με κάθε σεβασμό και συμπάθεια και όπως είπα θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ως Προεδρία αλλά εμείς δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα για σας. Εσείς πρέπει να δημιουργήσετε τη βάση να μπορέσετε να τα επιλύσετε. Δεν είναι καθόλου εύκολη η αντιμετώπιση και επίλυση αυτών των προβλημάτων ρεαλιστικά κιόλα εκτιμώντα το το λέω. Έχω κάθε σεβασμό για τι προσπάθειέ σα και τα όσα έχετε πετύχει μέχρι σήμερα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά, δεν επαρκούν. Πρέπει να προχωρήσετε παραπέρα, να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδο από πλευρά τη Βοσνία. Τώρα για τη Συρία. Για την ε, Λευκορωσία ήδη τοποθετήθηκα. Εδώ έχω κάτι άλλο μάλιστα. Λοιπόν, ειλικρινά πρέπει να πω ότι πάντα, προσωπικά πάντα, υιοθετώ τη θέση να είμαι νυφάλιος και ήρεμος, να μην υπάρχει φόρτιση ε, ε, συναισθηματική όταν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα με αυτή την ε, κατάσταση που δημιουργήθηκε και αυτό το περίγυρο που όλα συγχέονται. Θα πρέπει να είμαστε το δυνατόν πιο υπεύθυνοι και να συζητούμε με τους στρατηγικούς εταίρους μας με ένα επαγγελματικό τρόπο, νυφάλιο τρόπο για να μπορέσουν να αποσαφινιστούν όλα αυτά. Ξεκίνησαν όλα αυτά. Τη Δευτέρα μια ομάδα συνήρθε και συζήτησε όλα αυτά τα θέματα σε αυτό το πολιτιακό επίπεδο. Έγινε αυτή η αρχική συνάντηση. Ας ευχηθούμε κάθε επιτυχία, διότι πρέπει να αποσαφινιστεί το τι έγινε σχετικά με αυτή την περίπτωση. Όχι μόνο να αποσαφηνίσουμε τι συνέβη, αλλά και να διασφαλίσουμε ότι και στο μέλλον δεν θα υπάρξουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διότι η προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα του ανθρώπου είναι αξίες που βρίσκονται στην καρδιά, στον πυρήνα των αξιών μας και των αρχών μας. Όλα αυτά όμως να υπονομευθούν και να ε, διαλυθούν και να είμαστε όμοιροι μιας τέτοιας κατάστασης ε, για αυτά τα θέματα για παράδειγμα η Ιρλανδική Προεδρία ήταν ικανή και κατάφερε να προχωρήσει. Ήταν τόσο δύσκολα αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντικά όμω για την οικονομία μα. Είναι σημαντικό να υπάρξουν εμπορικέ ρυθμίσει για τι εμπορικέ σχέσει παγκόσμια. Μπορεί κανεί, να, να είναι πολύ φιλόδοξο, ώστε να υπάρξουν νέε προδιαγραφέ, να βελτιωθούν οι οικονομίε μα, να αυξηθεί το ΑΕΠ κατά το, μισή μονάδα έστω αμφωτέρωθεν. Αυτό πρέπει να είναι μία από τι προτεραιότητε μα, Όχι ει όλων των άλλων προτεραιοτήτων και στόχων, αλλά να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση επαγγελματικά, ήρεμα, νυφάλια, χρησιμοποιώντας επαγγελματικούς διάβλους. Δυστυχώς λέτε δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο να επεξηγήσω όλα αυτά, πρέπει εδώ να επαρκεστώ και να σταματήσω, έτσι. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Και τώρα έναν άλλο γύρο 15 λεπτών για κάποιες άλλες ερωτήσεις, αν γίνεται να το κάνουμε. Ah, Egypt was Egypt. Uh, Egypt. I Yeah ο κύριος Παλέτσκης, μάλιστα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να πω, κύριε Υπουργέ, για την Λευκορωσία τοποθετηθήκατε και είπατε και αναφερθήκατε σε μια σημαντική πτυχή για τη Λιθουανία και το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερθήκατε στην ε, ε, οικοδόμηση, στη δημιουργία ενός νέου πυρηνικού αντιδραστήρα εκεί. Εχθές ακριβώς συζητήσαμε τα θέματα της Μπελαρούς, της Λευκορωσίας και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι όταν απελευθερώνονται, όταν και αν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε, θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε, προσπαθήσουμε τότε να ξαναρχίσουμε ένα πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Λευκορωσίας. Φυσικά δεν υπάρχουν εχέγγυα, δεν υπάρχουν εγγύσεις ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά πώς πιστεύετε εσείς ότι ένας τέτοιος διάλογος θα μπορούσε να διαμορφωθεί και τι θα μπορούσαμε. Εσείς παρακαλώ κύριε Τζεβέβιτς. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι βέβαιος. αν ε, υπάρχει ακριβώς αυτή η δυνατότητα, αλλά τρεις ε, ερωτήσεις. Ε, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε υπό πόσο δύσκολους όρους ε, καταλήξαμε σε αυτή την προσέγγιση σε σχέση με την Μολδαβία Έχετε κάποιες ιδέες από πλευρά σας τι θα μπορούσε να γίνει από πολιτικές προτάσεις για να υποστηριχθεί αυτή η κατεύθυνση και να σταλεί ένα σαφές μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ αυτής της κατεύθυνσης και για την Λευκορωσία, Μπελαρούς. Ποιες είναι οι απόψεις σας, ποιες είναι οι δικές σας θέσεις για αυτό το θέμα. Θα μπορούσαμε να προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα για την περαιτέρω απελευθέρωση υπό το καθεστώς Λουκασένκα και όσον αφορά και τους... Εστία. παρακαλώ. Δεν παρίσταται. Όχι, εντάξει. Εδώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για αυτά τα οποία αναφερθήκατε στη Βοσνία Ζεγοβίνα. Το γεγονό είναι ότι αυτή η πολιτική οδήγησε σε σχέση με την ε, ιδιαίτερη εστίαση όσον αφορά στην ε, Ρωσία και Τουρκία θα μπορούσαμε να αναμείνουμε από τη Λιθουανική Προεδρία να ακολουθήσει μια πιο ενεργό πολιτική έναντι της ε, Βοσνίας Εζεγοβίνης και ποιοι θα ήταν συγκεκριμένοι στόχοι της Προεδρίας σας. Όταν αναφερθήκατε στη Σερβία τοποθετηθήκατε λέγοντας ότι υπάρχει ένας πολύ φιλόδοξος στόχος της έναρξης των διαπραγματεύσεων για τους Σέρβους πριν από τον Ιανουάριο. Τι θα λέγατε για τη, Σερβία, για τη Βοσνία Εζεγοβίνη, ποιες θα ήταν Uh, uh, Δεν αναφερθήκατε καθόλου, Υπουργέ, στις σχέσεις με την Ρωσία. Υπάρχει Ρωσία ακόμα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η Προεδρία σας ε, πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει τις ε, διαπραγματεύσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία κυρίως όσον αφορά την διμερή ε, συμφωνία. Αλλά και μην ξεχνάμε και την σύσταση που υιοθέτησε πέρυσι του, το Κοινοβούλιο. Επίσης ε, κάποια μέλη μας ε, συνυπέγραψαν μια επιστολή που σας στάλει και διαρωτώ με το θέμα αυτό θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις δεν απαντήθηκαν πλήρως, θα επανέλθουμε. Για την Αίγυπτο εξήγησα την κατάσταση, την ανησυχία μου για, τον, για την κατάσταση που επικρατεί και τη χρήση της βίας. Πιστεύω ότι ένα ε, δημοκρατικά εκλεγμένο καθεστώς δεν μπορεί να καθαιρεθεί από την στρατιωτική βία. Ε, ε, ούτως ή άλλως ε, δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την κατάσταση ούτε θα πρέπει να βιαστούμε να, κάνουμε, να επικυρώσουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί είναι διαφορά τώρα όσον αφορά την αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και, στην, και στο Συμβούλιο όσον αφορά την ε, τις εταιρικές σχέσεις ε, με την Ανατολική Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαχωρισμός. Ε, δεν παραπονούμε καθόλου. Υπάρχει συνεργασία και με την, με κυρία Άστον και με τον κύριο Φίλε. Οι πληροφορίες είναι ε, ικανοποιητικές η σύνοδος κορυφής του Βίλνιους δεν είναι του Βίλνιους, είναι στο Βίλνιους. Επομένως ε, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Τώρα για την Λευκορωσία, τι άλλο να πω. Είμαι υπέρ της δέσμευσης και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν πρέπει να χτίζουμε τύχη, πρέπει να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, διότι έτσι επηρεάζει. Και μία πρόσφατη απόφαση να, από τον Υπουργό Μακέιν. Είναι ακριβώς αυτό για, την, για τον κατάλογο, για την κατάργηση του καταλόγου. Ε, και αυτό είπα και στις, στο καθεστώς, ε, στην κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Δεν είναι κάτι καλύτερο ή χειρότερο. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κάποια βελτίωση. Είναι ένα κανάλι επικοινωνίας ε, το οποίο θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Και αν ο Υπουργό έρθει, τι θα πει ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να ε, ε, συζητήσει μαζί μας επικοδομητικά. Και αυτό θα είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον. Και μετά την ε, συνάντηση τα πράγματα θα είναι πιο ενδιαφέροντα και ελπίζουμε ότι θα προσεγγίσουν περισσότερο τον ευρωπαϊκό τρόπο σκέψη. Μην περιμένετε να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη τα πράγματα. Η δέσμευση είναι κάτι το θετικό. Για την Μολδαβία να σα πω, σας είπα ότι έχουν κάνει πολλά πράγματα. Επιλύθηκε το θέμα της κρίσης. Αντιμετωπίζουν βέβαια πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε να τους προσφέρουμε αυτά τα οποία είναι αναμενόμενα, δηλαδή να ξεκινήσουμε μια συμφωνία συνεργασίας, σύνδεσης, ε, όλες, όλα οι απαραίτητοι πόροι και γραφειοκρατικοί ακόμα να χρησιμοποιηθούν, διότι το έχουν κάνει, ίσως να τους δώσουμε μια δωρεάν βίζα για να έρθουν στις ε, συζητήσεις ε, και τους δίνουμε και ένα επιχείρημα προς, τον, προς τους τους πολίτες τους ε, ότι κάτι έχουν κάνει, κάτι έχουν πετύχει και αυτοί. Λοιπόν, για την Φωσνία, ειλικρινά δεν μπορώ να πω τίποτε παραπάνω. Να επαναλάβω ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να ασχοληθούν τώρα με την εφαρμογή ε, ε, της Ευρωπαϊκής Απόφασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα θέματα της διακριτικής μεταχείρισης πρέπει κάτι να κάνουν, δηλαδή πρέπει να κάνουν κάποια απτά βήματα, να μην μιλάμε θεωρητικά και να λέμε ότι α, πρέπει να ε, βελτιώσετε κάποια πράγματα, πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι μπορεί να γίνει. Επίσης, ε, η μία ε, να υπάρχουν κάποια, να γίνουν κάποια εφικτά βήματα και όσον αφορά τη συμφωνία σύνδεσης ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, για την ε, Ρωσία, Κριστίνα, δεν αναφέρθηκα γιατί δεν ε, ρωτήσατε. Καταρχάς, ε, η Ρωσία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα ε, συνεργασίας. Α, ο κύριος Μπρόκ, που είναι ο κύριος Μπρόκ, άλλαξε. Μπερδεύτηκα. Είπα κάτι, είπα κάτι κακό, γι' αυτό έφυγε. Ζητώ συγγνώμη. Θα πρέπει να εξηγήσω ότι ο κύριος Μπροκ ζητάει συγγνώμη, αλλά ε, πρέπει να πάει στην Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ τώρα. Και ζητώ συγγνώμη που σας διέκουσα. Λοιπόν, για την Ρωσία. Είμαστε στην διαδικασία επίτευξης αυτής της νέας συμφωνίας. Μπορώ να σας πω ότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι καινούριο, το reset δεν σημαίνει delete, γιατί ή το ένα ή το άλλο πρέπει να πατάμε και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Δηλαδή ε, πρέπει να γίνεται μια προσαρμογή. Δεν, η προσαρμογή δεν σημαίνει και κατάργηση και στην, ε, στον ΠΟΕ έχουν ληφθεί αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ε, δεν πρέπει να υπάρχει μια αρνητική στάση απέναντι στη Ρωσία. Καμιά φορά είμαστε, ε, συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε κλειστοφοβία, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν συνάντησα τον Λαυρόφ, ε, τρεις φορές έχουμε συναντηθεί μέσα σε ένα εξάμεινο και έχουμε ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις. Ε, υπάρχουν ε, βέβαια και θέματα αρνητικής, αρνητικά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Και όντως υπάρχουν αυτά τα θέματα, όμως αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θετικά σημεία και να κάνουμε κάτι για τα θετικά σημεία. Όλο αυτό το πράγμα θα πρέπει να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να διαγράψουμε τα αρνητικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια θετική προσέγγιση. Δεν θα πρέπει επίσης να επιτρέψουμε μια, την πρόσβαση από την πίσω πόρτα. Ε, ε, το καθεστώς για, τις, ε, για, την, για τη βίζα. Οι Ουκρανοί ίσως περάσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας περιελευθερωποίησης της βίζα αν πετύχουν αλλά δεν μπορούμε να χορηγούμε ε, δωρεάν βίζα για πολιτικούς λόγους. Πρέπει να ε, λειτουργούμε με βάση κάποια κριτήρια χρονικά ή αποτελέσματος. και όχι αναγκαστικά πιο γρήγορα από ό,τι απαραίτητα. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει το θέμα να αφορά τα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε και όχι απλώς και μόνο χρονικούς περιορισμούς ή όρια. Επίσης, ένα άλλο παράδειγμα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις ε, και άρθρα στην εφημερίδα, παραδείγματο χάρη, για το τρίτο πακέτο το ενεργειακό. Δεν είναι δικό μας θέμα, αλλά είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Και είχαμε πει ότι έπρεπε να το σταματήσουν, να σταματήσουν, διότι αλλιώ δεν θα ε, ε, μπορούσαμε να συνεργαστούμε, να συζητήσουμε μαζί τους. Αυτό δεν ισχύει, διότι έχουν δοθεί εξεγήσει. Δεν είναι η εθνική θέση της Λιθουανίας, είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θεωρούμε ότι η Ρωσία Ρωσία είναι ένας μεγάλος εμπορικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να έχουμε σχέσεις, αλλά εάν η Ρωσία θέλει να ε, παίξει ρόλο στην, ε, στην κοινοτική αγορά, πρέπει να παίξει με τους συγκεκριμένους κανόνες. Και στην ενεργειακή αγορά ισχύει το ίδιο. Επομένως, θα πρέπει ε, αυτή την, αυτούς τους κανόνες ε, να τους σεβαστούν. Και αυτό δεν είναι θέμα ε, τετελεσμένου. Δεν, ε, δεν τους επιβάλλουμε και δεν τους υπαγορεύουμε τι πρέπει να κάνουν. Είναι συγκεκριμένοι κανόνες. Το Μαγνίσκι, αναφερθήκατε στην υπόθεση Μαγνίσκι. Σαν Προεδρία θα προσπαθήσουμε να είμαστε αμερόληπτοι δεν θα ε, το θίξουμε εμείς, αλλά δεν θα το σταματήσουμε κιόλας. Υπάρχουν κάποιες συμβολικές υποθέσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν μεγάλες ε, ε, διαφορές στην αντιμετώπιση του κράτους δικαίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ρωσία. Υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να το κρύψουμε ή να το εξαφανίσουμε. Τώρα υπάρχουν οι κυρώσει. Οι κυρώσεις όμως είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Πρέπει να το χρησιμοποιούμε σαν τελευταία δυνατότητα. Πρέπει όμως όλα αυτά να συζητηθούν προσεκτικά και να δούμε αν τι μπορεί να γίνει κάτι. Τέλος πάντων, οι σχέσεις προχωρούν, εξελίσσονται. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε συνεπείς στη θέση μας και ελπίζουμε ότι θα ε, υπάρχει κάποια επιτυχία. Τώρα, στο τέλος, τώρα για τους πολιτικούς φυλακισμένους στην Λευκορωσία. Πρέπει να σας πω ευθύ εξ αρχής ότι όλα όσα, για μιλάμε, για δεσμεύσει, για κανάλια επικοινωνία, δεν πρέπει να γίνουν ει βάρο των πολιτικών ε, φυλακισμένων. Πρέπει να απελευθερωθούν. Δεν είναι και τόσο πολύ, είναι εφικτό αυτό. Θα πρέπει να πείσουμε τις αρχέ ότι μπορούν να, άρουν αυτό το εμπόδιο. Και με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουν οι δυνατότητες για ε, ενδεχόμενη συμμετοχή τους στο, στη Σύνοδο. Δεν λέω με πόσο θα παραστούν, αυτά θα τα συζητηθούν μετά την Υπουργική του Βίλνιους. Αλλά ε, ε, γίνεται αυτό και είναι θέμα ε, της πολιτικής μας. Το θέμα των φυλακισμένων για πολιτικούς λόγους πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να απελευθερωθούν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας, για, την, ε, τα όσα μας είπατε. Ε, καλή επιτυχία και ελπίζω να σας ξαναδούμε.